Ολομέλεια έλαβε γνώση ότι σε ό,τι αφορά την κατεξοδότηση πράξη δεν θα πρέπει να, γίνει, ε, να εκφραστεί ένσταση από την, ε, Ευρωπαϊ... από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και αν δεν υπάρξουν κάποιες αντιρρήσεις ε, θα τηρηθεί το άρθρο 105 παράγραφος 6 και θα θεωρηθεί η σύσταση αποδεκτή και θα δημοσιοποιηθεί αύριο 18 Απριλίου.